Λοιπόν, ακούσατε τα τρία χτυπήματα με το σφυράκι, που είναι το σήμα ότι μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την πρωινή μας συνεδρία. Ελπίζω να έχετε φέρει μαζί σας τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Να σας καλωσορίσω όλους θερμότατα. Πριν από λίγο οι συντονιστές ε, συνεδρίασαν με τον Υπουργό Γεωργίας της Βουλγαρίας που εγκαινιάζει την Προεδρία αυτό το εξάμεινο. Ένα κανονική συνεδρία των συντονιστών θα γίνει λίγο πριν το μεσημέρι. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες λοιπόν με πρώτο θέμα τις προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα της μελισσοκομείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Έρντος είναι ο εισηγητής μας. Και από ό,τι θυμάστε κατατέθηκαν γύρω σε 400 τροπολογίε και συμβαστικέ και η Επιτροπή έμβη γνωμοδότηση, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο εισηγητής που είναι και πλέον αρμόδιος. Έχετε το λόγο κύριε Έρντος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω ξεκινώντας να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και όλες τις πολιτικές ομάδες για τη βοήθεια που μου προσέφεραν. Τους και ηγητές και βέβαια το προσωπικό τους. Έχω δεχθεί κάποιες τροπολογίες. Νομίζω ότι πια έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η έκθεση έχει πάρει μια μορφή αποδεκτή για όλους. Έχουμε 39 συνολικά ε, συμβαστικές τροπολογίες, 35 χωριστές. Ε, περιμένουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας, αγρότες από την Αυστρία, μετά από πρόσκληση του κυρίου Βάιτ. Καλώς ήρθατε εκ μέρου του Πρόεδρου και ολόκληρη επιτροπή. Φτάσατε βέβαια σε μια τεχνική διαδικασία της ψηφοφορία, αλλά για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, που είναι η Ευρωπαϊκή Μελισσοκομεία. Τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε θα τι ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, τις υπόλοιπες τη της Ε, παρακολουθείτε τους συντονιστές σας. Πρώτη συμβαστική τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνούμε στην τρίτη συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τρίτη συμβαστική τροπολογία, παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία για την πέμπτη συμβαστική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 268. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 268. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 239. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 7α, τη συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. έχετε ε, ότι τη σημείωση ότι ψηφίζετε με την συμβαστική F. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 9α συμβαστική τροπολογία. Άρχεται ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 9α. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 39 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 378 παρακαλώ τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10, ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία τη συμβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία συμβαστική 13, τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική, μάλλον στην τροπολογία 40 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 40 της ΕΜΒΙ. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Υπάρχει ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστές, παρακαλώ. Εντάξει τώρα. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά η τροπολογία 40. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην 346-347 μαζί. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών 346 και 347. Είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 15 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 301. Ποιος είναι υπέρ κατά. 91 μάλλον είναι ο πρόεδρος. Ε, έλεγχος ηλεκτρονικός για την 301 λέει ο πρόεδρος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Οπότε η 13 της ΕΒ καταπίπτει. Και πάμε στην 397. Ποιος είναι υπέρ της 397. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία ηλεκτρονικός έλεγχος για την 391, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 391 και πάμε στην τροπολογία 18 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την τροπολογία 18 της ΕΜΒΙ άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αλλά στο ελέγξουμε καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 22 της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κύριε Ντες, ε, εγώ φταίω. Μέα κούλπα. Έκανα λάθος. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 17. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην συμβαστική τροπολογία 20. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 29 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ εγκρίνεται 287 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 422 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 423 ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 422 άρχεται η ψηφοφορία Μπορούμε να ξαναψηφίσουμε για τη 287. Ζητάει κάποιο. Η κυρία Νόιχλ συγκεκριμένα. Κανονικά είχαμε ψηφίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ζητάει η κυρία Νόιχλ. Α ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 287 πρώτα. Άρχεται ψηφοφορία για τη 287. Τέλος ψηφοφορίας. 422 τώρα ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 423. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 439 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 440. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. This is withdrawn. Oh, yes. And then, then last we vote for, for zero. No, no, false, because AV28 was Ach, okay. Yes, yes, yes, yes. Jest, dlatego, że wycofa, była przyjęta... Ναι, η 431 έχει καταπέσει. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε ούτε την 440. Πάμε στη συμβαστική κατευθείαν 29. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 29. Συμβαστική 29. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 450 και 451 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 450 και 351 ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Πάμε στην 452 και 453 μαζί πάλι. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 454 καταπίπτει λόγω έγκριση άλλων τροπολογιών και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 31 Άρχεται η ψηφοφορία. Α. Ε, επαναρχόμαστε στην 454, λέει ο πρόεδρος, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 31, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 32. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 476. Ποιος είναι υπέρ της 476. Υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 50 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ εγκρίνεται. 52 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ εγκρίνεται. 464 και 484 μαζί για την επανομοιότυπη υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο τροπολογίες 464 και 484. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 277. Ποιος είναι υπέρ της 277. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ. Α, μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά είπαμε τις συμβαστικές. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Πρόκειται για τροπολογία των Ταντά Νίκολσον Μαγκίνες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Α. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία Β. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 4 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική C και D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πάμε στην τροπολογία 42 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στις συμβαστικές τροπολογίες G και H. G και H, συμβαστικές τροπολογίες, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 81. Διανατάσσω στις χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία μη, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία νη, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 6 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ο, όμικρον. Ποιος είναι υπέρ. Ε, μάλλον ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία π. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στις συμβεστικές τροπολογίες Q και R. Άρχεται η ψηφοφορία για τις συμβαστικές τροπολογίες Q και R. Τέλος. Εγκρίνονται. Συμβαστικές τροπολογίες U και V. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται και πάμε στις συμβαστικές τροπολογίες XYZ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται και πάμε στις συμβαστικές τροπολογίες ΑΑ και ΑΒ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογία 160. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστικές τροπολογίες AC, A, AD και AE. Ψηφίζουμε τις τρεις συμβαστικές τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. AC, AD, AE. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία AF. Άρχεται η συμβαστική τροπολογία. Η ψηφοφορία, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία AFA νέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο ε, της έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. κύριε Ευρωβουλευτά, φοβήθηκα μήπως μας τελειώσει το αλφάβητο με τόσες συμβαστικές τροπολογίες με γράμματα αλφαβήτου. Ευτυχώς προλάβαμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. ...486 τροπολογίες είχαν κατατεθεί. Και αυτό δείχνει ότι χαίρει μεγάλου ενδιαφέροντος πλευρά των βουλευτών αυτή η έκθεση. Σα ευχαριστώ όλου όσοι λάβατε Μέρο Τώρα πιστεύω έχει γίνει ακόμη πιο συνεκτικό το κείμενο. Έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα μελήματα που εκφράστηκαν με τι τροπολογίε. Νομίζω ωστόσο ότι είναι πιο δομημένο το κείμενο και στις 28 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Ερντός. Καταφέρατε να συνοψίσετε αυτές τις πολυάριθμες τροπολογίες σχετικά λίγες συμβαστικές και καταφέραμε και ψηφίσαμε αισίως. Πάμε στο επόμενο θέμα, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται για γνωμοδότηση της κυρία Σοφία Ριμπέιρο ε, Πρόκειται για γνωμοδότηση επί της εκθέσεως πρωτοβουλίας της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αλλά να δώσω το λόγο καλύτερα στην κυρία Ριμπέρο που είναι η συγκέντρια της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα όλους τους πιο συγγητέ των πολιτικών ομάδων γιατί είχαμε πραγματικά εξαιρετική συνεργασία και καταφέραμε πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία επί των 7 συμβαστικών τροπολογιών που θα ψηφίσουμε και που καλύπτουν πάνω από τις μισές τροπολογίες που κατατέθηκαν. Ευχαριστώ και την ε, γραμματεία, ε, ε, τον κύριο Μπέζιλ Μάρτινς και τον γραμματέα από το ΕΛΚ. Νομίζω ότι έτσι διατρανώνουμε τη στεναρή θέση της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ της κοινή γεωργικής πολιτικής, υπέρ των αγροτών μας και υπέρ του γεωργικού προϋπολογισμού. Οι συμβαστικέ τροπολογίε καταδεικνύουν την τεράστια σημασία που έχει η ΚΑΠ για το γεωργικό εισόδημα και προσπαθούμε ε, όλο να έχουμε περισσότερε δράσει με λιγότερα κονδύλια και να καλύψουμε όλο και περισσότερε ανάγκε όπω η επιστηστική ασφάλεια, η καλή μεταχείριση των ζώων, αγαστέ περιβαλλοντικέ πρακτικέ και ούτω καθεξής. Θέλουμε ταυτόχρονα να έχουμε αγροεπιστηστικά προϊόντα μεγάλη ποιότητα σε προσιτέ τιμέ. Θέλουμε λοιπόν ένα γεωργικό προπολογισμό που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και θα έχει αρκετά ε, κονδύλια, αν όχι περισσότερα, τουλάχιστον στο παρόν επίπεδο. Ε, είμαστε υπέρ της ε, ισχύουσας διάρθρωσης ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες και ε, είμαστε κατά της, της απόπειρας επανεθνικοποίησης της κοινής γεωργικής πολιτικής που θέλουμε να παραμείνει κοινοτική. Και μάλιστα ενώψει ώψη αβεβαιότητας του Brexit εμείς ε, πιστεύουμε, ευελπιστούμε τουλάχιστον, ότι χρειαζόμαστε περισσότερη, ε, περισσότερες γεωρικές επενδύσεις ε, και μεγαλύτερη υποστήριξη της κοινή γεωρικής πολιτικής που θα είναι εγγύηση για την κοινωνική συνοχή στις ορεινές περιοχές, εξόχως απόκεντρες περιοχές, στην προστασία της οικογενειακής γεωργίας και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, αλλά και ε, τις ε, εξαγωγές, τις γεωρικές που αντιστοιχούν σε 130 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης θέλουμε να στηρίξουμε τους ε, χρήζοντες βοήθειας γεωργούς στις εξόχους απόκεντρες περιοχές. Γι' αυτό ταχθήκαμε υπέρ του προϋπολογισμού του ΠΟΣΕΙ. Είναι επίγουσα η ανάγκη δημιουργίας ενός κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών που δημιουργούν στρεβλώσει στη γεωργία. Μετά την ψηφοφορία Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα για να προασπίσουμε αυτές τις αρχές και αξίες και να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία, ανταποκρινόμενη στις ελπίδες των ψηφοφόρων μας. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε και εμείς να συμβάλλουμε στην ε, εδαφική και κοινωνική συνοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ πιο αντίξωε συνθήκες και αυτό να αντικατοπτριστεί και σε έναν επαρκή γεωργικό προπολογισμό. Ψηφίζουμε. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία επί της Συμβαστική τροπολογίας 1. Τέλος. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 9. Κατά απορρίπτεται, αλλά ή μάλλον απορρίπτεται όντως. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία 1α, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στις τροπολογίες 18 ε, ποιος είναι υπέρ της 18. Εγκρίνεται. 21 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 10 αρχή η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Πάμε στο 28 και 30. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. Τροπολογίες 29 και 31. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 2, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 38. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 44, υπέρ. Εγκρίνεται. 45, υπέρ. Εγκρίνεται. 47, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 49, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50, υπέρ εγκρίνεται 51 υπέρ εγκρίνεται 52 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 52 άρχεται ψηφοφορία Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Πάμε στην 57. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Κατά. Απερίφθη. 62 υπέρ, κατά. 66 υπέρ κατά. Απερίφθη 69 υπέρ κατά. Συμβαστική τροπολογία 4 άρχεται η ψηφοφορία. Otwieram głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 22, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ της 22, εγκρίνεται. Ή μάλλον... Πάμε στην τροπολογία 72. Ποιος είναι υπέρ, 72-82 μαζί, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία για τις 72 και 82. Τέλος. Εγκρίνεται. 78. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Εγκρίνεται. 83 συγγνώμη, παραλείψαμε την 75. Ποιο είναι υπέρ της 75? Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην 78. Ποιο είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 79 του κύριου Σάνι. ποιο είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 83 Νταντά υπέρ, κατά και ταραμπέλα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85 και 86. Ή μάλλον πρώτα ηλεκτρονικός έλεγχος για την 83, άρχεται ψηφοφορία. Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 85 και 86. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται απορρίπτονται θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο όχι 87 ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 87 εγκρίνεται 88 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 89 υπέρ κατά απορρίπτεται 90 ένα. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 91, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 92, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 93, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 95 και 96 υπέρ. Εγκρίνονται. 97 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 102. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 104 του κύριου Μπούντε υπέρ. Εγκρίνεται. 107 Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 108 Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 110 Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στα 121. 121 και 125 είναι πανομοιότυπες. Ψηφίζουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 121 και 125. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 122. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 124 άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται, μάλλον ε, ε, τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 126 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. κυρία Μίλλορ είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα. Γιατί δεν ξέρουμε οι φιλελεύθεροι πώς ψήφισαν. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 7. Ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 131 υπέρ εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά απορρίπτεται 133 υπέρ κατά απορρίπτεται ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης με τις τροπολογίες άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά και ονομαστικά Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε θερμά την εισηγήτρια την κυρία Ριμπέρο. Πώς έλεγε το λόγο πάλι κυρία Ριμπέρο. Ορίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατί είναι πολύ σημαντική, ήταν πολύ σημαντική η ψηφοφορία ε, και διατράνωση της θέσης της Επιτροπής Γεωργίας. Ελπίζω τώρα ε, θα είναι αξίσου φιλόδοξη και θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να στηρίξει και να βοηθήσει τις, την Ευρωπαϊκή Γεωργία και τους Ευρωπαίους αγρότες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ριμπέρο. Ευχαριστούμε και τους και ηγητές ε, και τους ε, ε, συνεργάτες. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών που είναι κατ' ουσίαν αρμόδια θα γίνει 21 και 22 Φεβρουαρίου. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 7. Τη γνωμοδότηση του κυρίου Καπούτο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της ουσίας αρμόδια είναι Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, συντάκτης γνωμοδότης, όπως είπαμε, είναι ο κύριος Καπούτο, που θα μας ενημερώσει για το θέμα, τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδιών πόρων. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες, τους και ηγητές για την δουλειά και τη βοήθεια στο θέμα αυτό. Ένα θέμα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει το σύστημα των ιδιών πόρων. Η Επιτροπή Γεωργίας δίνει, ε, απαντώντας στις προτάσεις, ε, με τις προτάσεις μάλλον για τους ίδιους πόρους, δίνει μια αποτελεσματική και επιφασιστική απάντηση. Μάλιστα. Είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα και πολύ σημαντικό. Πάντα το βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Παίρνουμε συμβαστική τροπολογία Α. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία B. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία C. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 33. 43, συγγνώμη, 43. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 44. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Κύριε Ντέση, σηκώνετε παρακαλώ το χέρι σας. 45. Ποιος είναι υπέρ. 45 υπέρ, εγκρίνεται. 48 πίπτη, γιατί τη 44 την εγκρίναμε. Πάμε στη 49 και 50. Μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ της 52. Εγκρίνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 51. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται. Οπότε πάμε στην 39, υπέρ, κατά, απορρίπτεται και αυτή. Δεν χρειάζεται. Κατά τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 39. Άρχεται η ψηφοφορία. 39, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εντάξει, όντω υπήρχε μια μικρή διακύμαση. αλλά απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία ε, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 42. 42 είπα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται εδώ είχαμε καλύτερη διακύμαση. 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Εγκρίνεται. Και Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το, σύντομο, το σύνολο της γνωμοδότης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η αρμόδια Επιτροπή Προπολογισμού θα ψηφίσει στις 21 και 22 Φεβρουαρίου. Πώς θέλει ο εισηγητής το λόγο μετά το πέρας της ψηφοφορίας της νομοδοτησής του. Καπούτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία νομίζω επιβεβαιώνει τη δουλειά που έκανα στις συνεδριάσεις. Η Επιτροπή Γεωργίας, λοιπόν, έχει ένα εξαιρετικό έργο να παρουσιάσει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε και το επιβεβαιώνουμε. Ευχαριστούμε και εσάς και τους συνεργάτες σας κύριε Καπούτο. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσια διάταξης, τις περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση. Η συντάκτηρα της γνωμοδότησης είναι η κυρία Νταντσίλα και αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η κυρία Τζουφρίτα έχει την έκθεση της Επιτροπής Ρέγγι. Περνάμε στην ψηφοφορία κατευθείαν, εκτός ε, αν θέλει κάποιος το λόγο Δεν χρειάζεται, μας λέει ο συντονιστής ο κύριος Αντρία, να λάβει κανείς το λόγο. Καλή γνωμοδότηση και καλή έκθεση, γιατί είναι σημαντική η θέση της γεωργίας στις ειστερούσες περιοχές. εκείνη που η γεωργία ε, τη χάνει ανάγκης ιδιαίτερης προστασίας στις Περιοχέ με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Παρακαλώ διαβιβάστε τα συγχαρητήριά μα στην κυρία Νταντσίλα που απουσιάζει στην εισηγήτρια τη γνωμοδότηση για την αξιόλογη προσπάθειά τη. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία τώρα τη γνωμοδότηση. Ξεκινάμε από τη συμβαστική τροπολογία Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Εγκρίνεται. Και πάμε στην ε, τροπολογία 27. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 28 εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά. Εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε καλού κακού. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεν είπα, δεν το είπα εγώ. Τροπολογία 30. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία B. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική C. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 39 παρακαλώ του κυρίου Καπούτο και της κυρίας Νταντσίλα. Ποιος είναι υπέρ της 39, εγκρίνεται. 44, ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 44, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Λάθος έκανα. Πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Και εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 52. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 63 της κυρίας Νταντσίλα, της ηγήτριας. Υπέρ. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Εγκρίνεται. 66 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία της συμβαστικής τροπολογίας G. Και τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 71, άρχιτη ψηφοφορία. Ε, μάλλον, συγγνώμη, ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 79, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Και πάμε στη βασική τροπολογία H, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 8. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική τροπολογία I. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 17 εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί ονομαστικά. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση και ευχαριστούμε την κυρία Δαντσίλα, την Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε τους και οδησηγητές, τους συνεργάτες, τους αντικαταστάτες και περνάμε στο σημείο 9, το τελευταίο θέμα που ψηφίζουμε σήμερα το πρωί. Συντάκτρια της γνωμοδότης για την απαλλαγή του 2016 είναι η κυρία Κάριν Κάντεμπαχ. Παρακαλώ έχετε το λόγο για μια εισαγωγή και ενημέρωση. Δεν χρειάζεται, λέει η κυρία Κάντεμπαχ. Περνάμε κατευθείαν στη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 1. Τι γίνεται, δεν ανοίγει. άνοιξε. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αλλά στο ελέγξουμε καλού κακού. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. 11 λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη. 11 υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα λέει 11. Υπέρ. Ή μάλλον 15, 15. Ποιος είναι υπέρ της 15 του κυρίου Σάνι. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα 11. Φλάνναγκαν, Τόρες και Μαρτίνες. Ποιος είναι υπέρ της 11. Εγκρίνεται. 12 καταπίπτει. 13 καταπίπτει επίσης. 14. Νταντά. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 16. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 17. Άρχεται ψηφοφορία. Νόμιζα ότι η κυρία Μιλέρη ήταν υπέρ. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 19 τεχνική τροπολογία. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 23. 3. 23 υπέρ. Εγκρίνεται. 24 υπέρ εγκρίνεται 25 υπέρ εγκρίνεται 26 υπέρ εγκρίνεται 27 υπέρ εγκρίνεται 28 υπέρ εγκρίνεται 29 υπέρ εγκρίνεται 30 υπέρ εγκρίνεται 33 υπέρ εγκρίνεται κατά μάλλον Απορρίπτεται η 33. Ή θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 33. Τέλος ψηφοφορίας. Και όντως απορρίπτεται. 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ίδιο αποτέλεσμα απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία εννοείται. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Θα τη δώσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού που είναι αρμόδια κατ' και που θα ψηφίσει μάλλον το Μάρτιο. Ο κύριος Σνέκοφ, παρακαλώ. νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε αυτούς για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα μάλιστα να σας δώσω γι' αυτό ένα βαζάκι με μέλι από τη Βουλγαρία που παράγεται στα βουνά της χώρας είναι μοναδικό προϊόν και είναι και το πρώτο προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης από τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ευρωβουλευτά, το απόγευμα ε, θα έχουμε την ευκαιρία να εγκομιάσουμε τη βουλγαρική γεωργία γιατί θα έχουμε καλεσμένο τον ε, βούλγαρο Υπουργό Γεωργίας που ασκεί και την Προεδρία του Συμβουλίου Γεωργίας. Είναι ήδη 10 και 8, αλλά η συνεδρίση των συντονιστών ε, προβλέπεται και τις 11. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Μπορούν οι συντονιστές να ξεκινήσουν 11 παρατέταρτο αντί για 11 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Όχι. Καλώς, κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε και μεγάλο διάλειμμα. Εντάξει. Όχι, μόνο 5 λεπτά διάλειμμα και θα ξεκινήσουν αμέσως οι συντονιστές.